περιβάλλον. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη συνεργασία και καλή σας νύχτα. Να Υποθέτω πως όλοι για ύπνο θα πάμε. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, ευχές. Κυρία Κουεστχούτ. Θα ψηφίσουμε αύριο, θυμίζω, στις 12. Η συνεδρίαση αρχίζει αύριο στις 9. Η ημερήσια διάταξη είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λήξη συνεδριάσεως.